Okay. If members would take their seats, please. Καθίστε αν θέλετε παρακαλώ. Jean-Paul, you want the floor? Oui, madame, madame la présidente. Madame, la... Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι που εργαζόμαστε σε αυτή την αίθουσα μαζί με την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών, αλλά με εντυπωσιάζει ότι δεν υπάρχουν τα ονόματα των βουλευτών της Οικονομικής Επιτροπής ε, δεν υπάρχουν τα καρτελάκια μας. Έχουμε δικαίωμα να ψηφίσουμε ή όχι. Τα ονόματά μας είναι στην αίθουσα εκεί που θα ξαναγυρίσουμε σε μία ώρα, λέει η πρόεδρος. Και οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου δεν έχουν βρει κάποιο σύστημα με το οποίο να μεταφέρουν τα καρτελάκια. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ότι αν έχω δύο, όταν έχω δύο κόρες αγαπάω και τις δύο. Και ο Φρασό Ολάν δεν είπε ότι αν έχω δύο γυναίκες τις αγαπώ και τις δύο εξίσου βέβαια. Παρατηρεί κάποιος. Well, anyway, we're going to start Εντάξει, θα ξεκινήσουμε γιατί είναι 9 και 4. Δεν ξέρω αν είναι αρκετά μέλη εδώ ή όχι για τις ψηφοφορίες. Please, παρακαλώ. Νομίζω ότι έχουμε αναμείνει αρκετά για να έρθουν τα μέλη, είτε έχουν τα καρτελάκια τους είτε όχι. Παίρναμε πρώτα στην έγκριση μερικές διάταξη. Δεν βλέπω καμία αντίρρηση ή κάποια αίτηση για τροποποίηση, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Και το θέμα που μας ενδιαφέρει τώρα είναι η ψηφοφορία. Βάλτε τις κάρτες σας να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία, αν θέλετε. Ανοίγω την ψηφοφορία. Okay, we have technical problems that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 το σύστημα μας λέει ότι έχουμε τέσσερα μέλη του, των φιλελευθέρων της Άλντε πάνω από την ποσόστοση. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι δυνατό, ούτε δέσεις δεν είναι εδώ παρόντες. Who's Ποιοι είναι εδώ από την Άλντε, τέσσερα άτομα πράγματι. Three, four. Λοιπόν, κάτι δεν δουλεύει καλά στο σύστημα. Η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων έχει τέσσερα μέλη μόνη της. Καλά, δεν θα κάνουμε σήμερα ηλεκτρονικές ψηφοφορίες μάλλον. It's, look, it's saying we've got four Aldi members too many and we've only got five Aldi members here. Εδώ λέω ότι περισσεύουν τέσσερις από την Άλντε και έχουμε πέντε μονάχα παρόντες εδώ. Τι γίνεται. We've only got five in the room, so it's wrong. Normally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 Για πατήστε το κουμπί να δούμε τι θα βγει. Τώρα μου λέει ότι όλη η Επιτροπή είναι φιλελεύθερη. Λοιπόν, 61 κάρτες και 53 χτύπησαν, ε, πίεσαν το κουμπί, 54 πίεσαν το κουμπί τους, 61 είναι συνδεδεμένοι, 57 έχουν ψηφίσει, 58 59 Δύο ακόμα δεν έχουν ψηφίσει. Θα ψηφίσετε. Δύο δεν έχουν ψηφίσει. Κάποιοι ίσως δεν είναι στην ε, θέση τους. Με ενοχλεί ότι οι δύο κάρτες δεν λειτουργούν. Πάμε. Τροπολογία 11. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίντ Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 11 ζούρι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ για την 14 άρχεται Well, I'd like somebody... Oh, yeah, okay. Uh, that's 33 26 εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 15 υπέρ. Κατά Υπάρχει μια προφορική τροπολογία εδώ. Να έχουμε και τα ηλεκτρονικά χρήματα μετά τα κινητά τηλέφωνα. <clears throat> Με την προφορική αυτή τροποποίηση υπέρ κατά αποχές δεκτή 68 είναι συμβατή υπέρ κατά αποχές δεκτή 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε τη 16 παρακαλώ Uh, and that's carried 31. Εγκρίνεται 31-27, τροπολογία 70 υπέρ. Κατά. Απόχες απορρίπτεται. Συμβαστική A υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Απόχες δεκτή. 73 υπέρ. Κατά. Απόχες απορρίπτεται. Γιούρι 13 είναι ταυτόσιμη. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος άμα θέλετε. Εγκρίνεται 36 με 24 76 υπερ κατά αποχές θα την ελέγξουμε. Νομίζω ότι εγκρίνεται. «35-23» εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 γιούρι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για 15 γιούρι 28-31 απορρίπτεται. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 80 ψηφίζεται. Δεν ψηφίζεται. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 αποσύρθηκε. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ογδόντα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 93 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 93 παρακαλώ εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 γιουρί υπέρ κατά αποχές μπορούμε να την ελέγξουμε τη 18 άρχεται ψηφίσατε όλοι εγκρίνεται 34-25 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 με προφορική τροποποίηση απαλήφεται το τμήμα που αφορά τους εθνικούς νόμους με την προφορική τροποποίηση υπέρ υπέρ κατά αποχές δεκτή 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 εκπίπτει 110 υπέρ κατά αποχές δεκτή να την ελέγξουμε την 110 αν θέλετε όχι δεν χρειάζεται 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή 112 υπέρ κατά αποχές δεκτή 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή και οι άλλες δύο είναι ταυτόσιμες 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές εδώ έχουν αλλάξει οι πολιτικές ομάδες 120 ελέγχουμε ηλεκτρονικά ψηφίσατε όλοι 30-31 απορρίπτεται Συγγνώμη να ξαναελέξουμε την 120 γιατί ήταν τρεις ακόμα που θέλαν να ψηφίσουν. Ελέγχουμε και πάλι την 120. Γιατί η γραμματεία έκλεισε την ψηφοφορία προτού τους δώσω εντολή να το κάνουν. Ενώ κάποιοι προσπαθούν να ψηφίσουν. 120 την ξαναελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ίσως αλλάξει, αλλά εγώ προσπαθώ να είμαι ισοδίκαια. Άλλο ένα δεν έχει ψηφίσει. Καλά, αν δεν ψηφίσει θα την κλείνω την ψηφοφορία. Μα έχετε ανακοινώσει το αποτέλεσμα. Επομένω έχει κλείσει το θέμα. Λέει κυρία Ματιέ. Ναι, εξακολουθεί να έχει απορριφθεί η τροπολογία, οπότε δεν υπάρχει θέμα, λέει η πρόεδρος. Μα όταν ανακοινώνεται το αποτέλεσμα έχει τελειώσει. Δεν μπορείτε να ξαναψηφίσετε, το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Αν δεν πω ότι έχει τελειώσει η ψηφοφορία, μην την σταματάτε, μην την κλείνετε. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 121. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 122 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 122 Δύο ακόμη να ψηφίσετε, παρακαλώ. Ο ένας από τους δύο ψήφισε, εγκρίνεται. Πανομοιότυπες 33 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 123 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 124. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 125. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 127 Τρει ακόμη να ψηφίσουν, παρακαλώ. Δύο πέρα στις ψηφοφορίες, θα την κλείσουμε. Απορρίπτεται. 128. Υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε για την 128. 128. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Δύο ακόμη να ψηφίσουν. Ένα, κλείνει ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 32 προς 31. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 131 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 136. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 137. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 138. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 139 υπέρ, κατά, απόθέσει εγκρίνεται. 100 να ελέγξουμε για την 139. 3 ακόμη να ψηφίσουν παρακαλώ. Δύο, ένας, κλείνει η ψηφοφορία εγκρίνεται 36 προς 26 140 υπέρ κατά αποχές οι σοσιαλιστές δεν ψηφίζουν γι' αυτό θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά θα ελέγξουμε για την 140 Κλείνω την ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται 36 προς 26. 141 υπέρ. Όχι, έχει καταπέσει. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 143 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 144 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 145 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική ή ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2 υπέρ. Κατά. απόχέ Εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Με συγχωρείτε έχει, πέσει, έχει καταπέσει. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε για το 49. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 49. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 29 υπέρ 33 κατά. 50 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε για την 50. Πέρας. Εγκρίνεται με διαφορά. 6 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ έχουν καταπέσει. Και η 53. Η 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 55. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε για την 55. ψήφισαν άπαντες πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 36 προς 26. Μισό λεπτό. Συμβατή 56 υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε για το 56. Νομίζω ότι θα εγκρίθηκε, αλλά ας το δούμε. Δύο ακόμη ψηφίστε. Πέρας. Απορρίπτεται. 30 υπέρ, 32 κατά. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεβεπτά υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Γιούρι 3 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύε 8 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Δεύε 9 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές να ελέγξουμε για το 58. Δύο ακόμη να ψηφίσουν κάποιος που δεν είχε ψηφίσει πριν, ψηφίζει πρώτη φορά, πέρας της φοβοριας απορρίπτεται. Ντεβε 10, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Γιούρι 4, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 5 Εκαταπιπτή. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 Καταπιπτή. 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 6 Καταπίπτη. Γιούρι 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 κατά πίπτη ή 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά στο τροποποιημένο, για το τροποποιημένο κείμενο τελική ψηφοφορία Εψήψαν άπαντες πέρας της ψηφοφορίας 57 υπέρ, 5 κατά, μία αποχή. Και τώρα ηλεκτρονική ψηφοφορία για το κοινοβουλευτικό ψήφισμα. Εψήφισαν άπαντες δύο ακόμη. Παρακαλώ να ψηφίσουν. Κλείνω την ψηφοφορία. 56 υπέρ, 5 κατά, μία αποχή. Δεν θα ψηφίσουμε για τη διαπραγματευτική εντολή, διότι προφανώς θα περιμένουμε και αυτό θα γίνει με την πρόταση κομπάνιων τη συνοδευτική. Ε, ευχαριστώ όλους που ψηφίσατε. Τουλάχιστον εδώ τελειώσαμε από την πλευρά της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Οι εισηγητές θέλει κανείς να σχολιάσει. Ωραία.